Συνάδελφοι, καλησπέρα. Ελπίζω να περάσατε ωραίο Σαββατοκύριακο και να σα έλειψα. Περνάμε στην έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει την εγκρίνουμε ω έχει. Κύριε Κάμπ, καθίστε παρακαλώ. Ηρεμήστε. Σταματήστε να κάνετε πηγαδάκια με του συναδέλφου. Αρχίζει η συνεδρίαση. Με το πάσο σας, κύριε Βαντεγκάμπ. Δεν βιαζόμαστε. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3ης Δεκεμβρίου τα έχετε λάβει. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνονται. Και περνάμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Ευχαριστώ. Να σας ανακοινώσω ότι οι αποφάσεις έχουν λάβει οι συντονιστέ στη συνεδρίαση της 10 η Ιανουαρίου έχουν μοιραστεί σε αντίγραφα στην αίθουσα και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει ως τι 5.30 θα θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένε. Και απλώς να σα θυμίσω ότι λόγω χρονικής πίεσης, σοβαρής χρονική πίεσης, αποφασίσαμε ομοφόνο στην συνεδρία των συντονιστών να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία βάσει του άρθρου 50 του εσωτερικού κανονισμού για τα τρία νομοθετικά ντοσιέ που αφορούν τον Brexit. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο στο δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα τρία κείμενα θα δημοσιευθούν εγκαίρω στην επίσημη εφημερίδα ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε νομική αμφισημία. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητή θα πρέπει να υποβάλει τροπολογίε, εάν αυτέ είναι απαραίτητε, έω την Τετάρτη 23 του μήνα, δηλαδή σε δύο μέρε. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές ομάδες και οι σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να ε, συζητήσουν ω το δυνατόν πιο σύντομα με τον εισηγητή, γιατί μόνο ο εισηγητή μπορεί να υποβάλει τροπολογίε βάσει του άρθρου 50 του εσωτερικού κανονισμού. Την διαδικασία την γνωρίζετε πλέον, οπότε περνάμε σε ένα θέμα σοβαρότατο, σημαντικότατο και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο κύριος Σβόμποντα και η κυρία Χάταλα είναι εδώ για να το συζητήσουμε. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα συζητήσουμε για την πρόταση οδηγία που θα προβλέπει τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών τη ώρα καταργώντα την οδηγία 2084. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην εισηγήτρια και μετά στους κοιόδης εισηγητές και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και μετά θα, καλήσω, θα καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο για να ολοκληρώσουμε την εισηγητρία. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 28 Ιανουαρίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινούμε ευθύ αμέσως με την εισηγητριά μας, Η κυρία Ούλσκοφ δεν είναι εδώ. Οπότε θα την ε, αντικαταστήσει η κυρία Χέτ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν καταλαβαίνετε, βάλτε καλύτερα τα ακουστικά σας. Λοιπόν, όπως είπε η Πρόεδρος, εκπροσωπώ τη Μαϊτά Γουλσκοπ, η οποία ζητεί συγγνώμη που δεν κατάφερε να παραστεί σήμερα εδώ, για να σας παρουσιάσει την έκθεσή της για τον τερματισμό των εποχιακών αλλαγών της Αλλά δεδομένη της πολιτικής κατάστασης στη Σουηδία πρέπει να σας πω ότι έχουμε πλέον κυβέρνηση, δυστυχώ καθυστέρησε στο ταξίδι τη. Ε, και ελπίζει, είναι στις Βρυξέλλες και ελπίζει να φτάσει εδώ εγκαίρως για το συζήτηση που θα έχουμε αμέσως μετά. Είναι υπέρ του τερματισμού των εποχιακών αλλαγών της ώρας η συγγήτρια. Ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκαν οι αλλαγές για τη θερινή ώρα ε, δεν ισχύει πια, διότι δεν χρειάζεται πλέον να εξοικονομούμε με αυτόν τον τρόπο ενέργεια. Δεν υπάρχουν πλέον οι ίδιες επιπτώσεις όπως παλαιότερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές. Παρ' αυτά η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ένα μια συντονισμένη προσέγγιση για τις μεταφορές, την αγορά εργασίας και γι' αυτό θα πρέπει για λόγους εσωτερικής αγοράς ε, να δώσουμε επαρκή χρόνο, ιδίως στον κλάδο των μεταφορών και να υπάρχει προβλεψιμότητα μακροπρόθεσμη, ώστε οι όποιες αλλαγές γίνουν να μην επηρεάσουν αρνητικά τους καταναλωτές μας. Ο κλάδος των μεταφορών θα είναι κατά πάσα πιθανότητα εκείνος που θα επηρεαστεί περισσότερο από όλους τους άλλους. Σκεφτείτε μόνο τις πτήσεις. 13.000 πτήσεις ε, ε, πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει μια τέτοια αλλαγή σημαντικές ε, επιπτώσεις στον κλάδο των μεταφορών. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο κλάδος που θα επηρεαστεί. Ε, των οδικών μεταφορών δηλαδή, ε, ο κλάδος της αεροπορίας είναι εκείνος που χρειάζεται τον περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στις όποιες αλλαγές και γι' αυτό η συγγήτρια προτείνει να υπάρξουν 18 μήνες μεταβατική περίοδος. Αν, κάποιος θέλει, αν κάποιο κράτος μέλος θέλει δε να αλλάξει τις, τους κανόνες του, τους εσωτερικούς, θα πρέπει να το ανακοινώσει 18 μήνες εκ των προτέρων. Και αυτό θα ήταν προτιμητέο παρά να ορίσει η οδηγία η Κομισιόν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντιθέτως λοιπόν η εισηγήτρια προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή να τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια από τη στιγμή της κοινοποίηση. Η εισηγήτρια καλεί παρόλα αυτά να εγκριθεί η οδηγία φέτος, να θεσπιστούν και να δημιουργηθούν δίκτυα ώστε να υπάρξει επαρκής και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ εκείνων που προτίθενται να αλλάξουν τους κανα... κανόνες τους. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια τυποποίηση, μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Να μην καταλήξουμε δηλαδή σε ένα τεράστιο μοσαϊκό με διαφορετικές χώρες να έχουν διαφορετικές διευθετήσεις για την ώρα τους. Και συμπερασματικά ε, η συγγήτρια θέλει να ευχαριστήσει όλους τους κοιόδης, οι εισηγητές για τη συνεργασία κτλ. Ε, ευχαριστούμε κυρία Χέτ. Κύριε Σφόποντα, πρόσωπο των πολιτικών ομάδων τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πρόταση που μας υπέβαλε, την οποία χαιρετίζω και και εγώ ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε η εκπρόσωπός της. Εδώ βέβαια έχω διπλή ιδιότητα, είμαι και σκιώδης εισηγητής, αλλά είμαι και εισηγητής για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για αυτό το θέμα. Οπότε, Η άποψή μου έχει διπλή βαρύτητα, γι' αυτό θα υποβάλω τροπολογίες. ώστε αυτού του είδους η πρωτοβουλία Αυτό το είδους η πρωτοβουλία για τα θέματα της υγείας κυρίως αλλά και των μεταφορών σε αυτά θα έχει τις μεγαλύτερε επιπτώσεις, θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που θα διοργανώσουμε και αυτό το μίνι σεμινάριο, τη συζήτηση, για να φωτίσουμε καλύτερα το όλο θέμα ώστε να μην ξεχνάμε ότι κυρίως η υγεία επηρεάζεται από αυτές τις αποφάσεις και για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να σταματήσουμε να αλλάζουμε τα ωράρια από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Αυτού του είδους τα επιχειρήματα είναι σημαντικά γιατί ακριβώς άπτονται της προστασία της υγείας. Θα πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση για το θέμα αυτό, ώστε να μην θέσουμε αμφιβόλο και την ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Σβαμποντό. κύριε Λουτόφσκι. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Όλσκοφ για την ε, εκπόνηση αυτής της έκθεσης Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις προτάσεις τροπολογιών. Προβλέπονται δύο χρόνια μεταβατικής περίοδου πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας και την κατάργηση των αλλαγών. Είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστούν καταλήλως όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Βάσει της πρότασης της εισηγήτριας, πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που με τη σειρά της θα πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα για τα θέματα αυτά και να ελέγχει κατά πόσο οι αρμοδότητες που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη εκπληρώνονται. Δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν για την ε, διεξαγωγή και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις της και δεν έχει εκπονήσει η μελέτη αντικτύπου της πρότασης αυτής. Έχουμε λοιπόν την προσδοκία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορέσει να εκπονήσει τη μελέτη αντικτύπου για την οδηγία αυτή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ζουσλοτόφσκι. Κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Bonjour, muchas gracias a todos. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Συζητήσαμε και εδώ στην Επιτροπή αυτή την πρόταση που ξεκίνησε από την Επιτροπή Μεταφορών, αλλά αντιαποκρίνεται σε μια πρωτοβουλία των πολιτών. Ο σημαντικό αριθμό ε, ανθρώπων που συμμετείχε σε αυτή τη διαβούλευση από πλευρά των κρατών μελών μας ε, έκανε να ασχοληθούμε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εργασία της και υπάρχουν δύο τουλάχιστον πτυχές που θα ήθελα να τονίσω πρώτον η ανάγκη εφόσον καταργηθούν οι αλλαγές ωραρίου, να υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μην υπάρξει αντίκτυπος και συνέπειες και κυρίως ε, να μην ε, επηρεαστεί ο τομέας των μεταφορών με τον οποίο ασχολούμαστε εμείς. Επίσης, ε, κατά δεύτερο λόγο, υπόθηκε ότι θα πρέπει το κάθε κράτος να αποφασίσει ποιο ωράριο θα ακολουθεί υπάρχουν και κάποιες επιτυχίες που δεν είναι πολύ σαφείς και εν πάση περιπτώσει με τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Στις τροπολογίες της ε, δεν φαίνεται, δεν ορίζεται ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται οι αλλαγές και οι προτάσεις να προταθούν από τα κράτη-μέλη. Ωστόσο δεν ε, Αναφέρεται κάπου ρητά ο συντονιστικός ρόλος που φαντάζομαι θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτές τις αλλαγές. Ε, δεύτερον, πιστεύω πως θα είναι καλύτερο να έχουμε περισσότερο χρόνο για να το, να το αλλάξουμε, αλλά να το κάνουμε όλοι μαζί. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει μεταξύ μας να ορίσουμε μεταξύ όλων ε, κάποια ημερομηνία ε, συγκεκριμένη ώστε να μπορέσουμε όλοι να εφαρμόσουμε την αλλαγή αυτή γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους ε, τομείς και αλλά και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου που θα γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Το Συμβούλιο ΔΕ, από ό,τι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, φαίνεται να μην θέλει να προχωρήσει ε, σε αυτή την ε, υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου ή, εν πάση περιπτώσει, η υπεύθυνη των κρατών μελών για αυτό το θέμα. Για να μην ε, έχουμε προβλήματα όταν θα ληφθεί η απόφαση. Τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν καλό θα είναι να προχωρήσουμε σε αυτή την έκθεση αλλά να δούμε και ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου που δεν ξέρω αν τώρα η Κομισιόν μπορεί να μας ενημερώσει ή αν θα το αφήσουμε για την επόμενη ε, θητεία. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Νταλούντε, έχετε το λόγο. Η πρόταση να, αλλα... να σταματήσουν οι αλλαγές ωραρίου, να εγκαταλείψουμε τώρα αυτήν την τακτική αλλαγή ωραρίου θα είναι θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα για το διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο θα ωφεληθεί από την πάυση αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αυτά τα ωφέλη θα είναι δυνατά μόνο όταν θα συντονιστούν τα κράτη-μέλη καταλήλως και αυτό κάπως μας ανησυχεί όσον αφορά τις ε, εξελίξεις. Γιατί προτείνεται τα κράτη-μέλη να λάβουν μεμονωμένα τις αποφάσεις αυτές. Αν η Κομισιόν έχει λάβει εντολή διαπραγματευτική για να συντονίσει τα κράτη-μέλη, δεν είναι σίγουρο ότι θα ε, ταιριάξουν οι αλλαγές. Το κόστος ε, μη συντονισμένων αλλαγών θα είναι ψηλότερο από τις ισχύουσες ε, ε, μέχρι τώρα αλλαγές ε, στο χειμερινό και στο θερινό ωράριο. Γι' αυτό και παροτρύνω όλους να εργαστούμε προς την εναρμόνιση από πλευρά των κρατών μέλλον. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαντεκάμπ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε θα πρέπει να πω ότι ο συντονιστής οι μεταφορές στις μεταφορές τους τελευταίους μήνες παρακολούθησα όσο γινόταν καλύτερα αυτή τη διαδικασία και πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την έκθεση του Σκιώδη Βόμποντα και των βοηθών του, αλλά προσωπικά ε, δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι υπέρ του συστήματος που ισχύει. Αν δω αν δει κανεί μάλλον το τι κάνουν οι αθλητικοί όμιλοι στις κάτω χώρες, είναι δυσαρεστημένοι από, την, από το θερινό ωράριο. Μπορούν να ασκούν τις αθλητικές δραστηριότητε ε, ικανοποιητικά και επίσης ε, να ε, εκμεταλλευτούν την μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας, βεβαίως το πάνελ των εμπειρογνωμόνων θα μας ενημερώσει. Πότε κατάλαβα, 5 εκατομμύρια κόσμος ανταποκρίθηκε στη διαβούλευση. Οι υπόλοιποι 485 εκατομμύρια γιατί δεν έλαβαν θέση. Αυτό σημαίνει πως η πλειοψηφία που δεν έλαβε θέση στη διαβούλευση παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Τι ακριβώς συμβαίνει. ή μήπως δεν το απασχολεί. Από τον συνάδελφο Σβόμποντα και τώρα και από την ε, συνάδελφο που αντικατέστησε την εισηγήτρια ακούμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μία ευρωπαϊκή ώρα. Βεβαίως ε, με τις διάφορες ε, τα διάφορα ωράρια λόγω της γεωγραφικής θέσης. Αυτό όμως δεν έχει επιρροή στην εσωτερική αγορά. Στις κάτω χώρες αν χρειαστεί να το κάνουμε αυτό, εμείς θα θέλαμε να διατηρήσουμε το χειμερινό ωράριο. Και συμφωνώ με την κυρία Μπιλμπάου, γιατί άκουσα και εγώ ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να κινηθεί. Όμως, γιατί οι δέσμοι περικινητικότητας έχουν ε, φτάσει σε κάποια κοινή θέση. Ας μην αρχίσουμε τώρα με τη συζήτηση του πακέτου κινητικότητας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για, τις, για τα ωράρια. Από ό,τι κατάλαβα και ο κύριος Ρικέ και εσείς ε, είσαστε μηχανόβοι. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το συζητάμε. Ε, με μεγάλο ταρατατζούμ ο κύριος Γιούγκερ πέρσι ανακοίνωσε ότι θα καταργηθεί η αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη και πλέον γίνονται σοβαρές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τι να πω, όδινεν όρος και έτεκεν μην. Πρέπει να σας πω δε ότι ούτε ο τίτλος της ε, οδηγίας δεν είναι σωστός. Θα έπρεπε να είναι άλλος ο τίτλος, διότι δεν μιλάμε απλά για μια αλλαγή από τη θερινή προς τη χειμερινή ώρα. Αντιθέτως, όπως βλέπετε και στην έκθεση της ε, εισηγήτριας, στην πραγματικότητα ε, πρόκειται για μια αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, αλλά μετά από δύο χρόνια. Άρα δεν ισχύει ο τίτλος, διότι η αλλαγή θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα και ε, στη διάρκεια αυτών των επόμενων δύο ετών. Οπότε αναρωτιέμαι τι ακριβώς συζητάμε εδώ σήμερα. Αλλαγέ στην ώρα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης υπάρχουν, αλλά ακόμα και αν ακολουθήσουμε τη γραμμή της εισηγήτριας, ε, μπορεί να καταλήξουμε στο τέλος η Γερμανία να έχει άλλο σύστημα για την ώρα, άλλο σύστημα η Ολλανδία, άλλο σύστημα το Βέλγιο. Ε, τόσο σκόπος αξίζει να γίνει. Μήπως, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε μια συζήτηση γύρω από το φύλλο των αγγέλων, μήπως τελικά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία όλο αυτό το θέμα, μήπως τελικά τζάμπα εργαζόμαστε και συζητάμε τόσο καιρό για αυτό το θέμα. Ιδίω δε, δηλαδή, αν ε, θεσπιστεί και μια μεταβατική περίοδο δύο ετών, μήπω εν τέλει το μόνο που κάνουμε τόσο καιρό είναι να σπαταλάμε χρόνο και χρήμα, Μήπω έχουμε και καλύτερα πράγματα να κάνουμε, Μήπω του εμπειρογνώμονε που έχουμε καλέσει σήμερα θα μπορούσαμε να του είχαμε καλέσει και για σοβαρότερα θέματα. Ευχαριστούμε κύριε Φαντάλεν. Είστε σε φόρμα. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Αν και γενικά συμφωνώ με τον Πέτρο Βαντάλεν, ε, σε αυτό το θέμα έχω διαφορετική άποψη. Κάθε άλλο παρά φάρσα είναι το θέμα αυτό. Εγώ ασχολούμαι με το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται υπέρ τη κατάργηση τη θερινή ώρα, η οποία θεσπίστηκε για να εξοικονομηθεί ενέργεια, για να αποφευθούν ατυχήματα τις βραδινέ ώρες. όμω τελικά διαπιστώθηκε ότι ο στόχο αυτό δεν επετεύχθη με την αλλαγή τη ώρα. Αντιθέτω, για τι εσωτερικέ μεταφορέ υπήρχαν πολλέ φορέ και προβλήματα με τα οδικά προγράμματα, με τα χρονολόγια προγράμματα. Υπήρξαν δε και πολλές επιπτώσεις αρνητικές στην υγεία. Διαπιστώθηκε ότι η κατάθλιψη ε, πήρε την άνοδο ε, στην, ε, στην Ευρώπη, ακόμη και αυτοκτονίες διαπιστώθηκαν, τα παιδιά έχουν χειρότερες σχολικές επιδόσεις, οπότε υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα να καταργηθεί αυτή η αλλαγή της θερινής ώρας, αφού οι διακηρυγμένοι στόχοι που οδήγησαν στην αλλαγή δεν επετεύχθησαν. Λοιπόν, τώρα μπορεί και να ε, υπερβάλλω λίγο. Δεν λέω ότι τα, οι μαθητέ μα θα γίνουν οι καλύτεροι και οι Ευρωπαίοι θα γίνουν οι πιο υγιεί στον κόσμο. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να καταργηθεί η αλλαγή τη θερινή ώρα. Είχα μάλιστα κάποτε συζητήσει και με τον Επίτροπο Κάλλα μήπω θέλει μια τέτοια διαδικασία να, να την ξεκινήσει. Εκείνο μάλιστα, μάλιστα μάλλον μου είχε πει ότι η Παναγία μου είναι καυτή πατάτα αυτό το θέμα. Δεν το αγγίζουμε γιατί ε, το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να πούμε στις χώρες ότι καταργούμε την οδηγία. Δεν μπορούμε να τους πούμε τι ώρα θα έχουν. Στη Σοβιετική Ένωση ε, πρέπει να σας πω ότι κάποτε είχε θεσπιστεί η θερινή ώρα αλλά καταργήθηκε. Γιατί δεν επετέφθηκαν οι στόχοι. Γιατί πρέπει εμεί λοιπόν να φανούμε πιο χαζοί από ότι οι Σοβιετικοί. Φυσικά και θα ήταν ιδανικό να έχουμε την ίδια ώρα σε ολόκληρη την, ε, την Ευρώπη, αλλά ε, αυτό ε, δεν επιτυχάνεται από τα πάνω. Να φανταστείτε ότι ε, όταν θεσπίστηκε στην Ευρώπη η θερινή ώρα, στην Ελβετία δεν θέλαν να κάνουν σχετική αλλαγή. Όμως την κάναν ακριβώς για να ακολουθήσουν τους γείτονές τους, για να μην υπάρξουν οικονομικά μειονεκτήματα για τη χώρα. Η γνώμη μου λοιπόν είναι να καταργήσουμε τη θερινή ώρα, να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση, στη χειμερινή ώρα, δηλαδή την κανονική ώρα με άλλα λόγια, την τυπική ώρα, διότι αυτό έχει διαπιστωθεί από τις έρευνας και μάλιστα έχουν δοθεί μέχρι και βραβεία Νόμπελ σε ε, γιατρούς οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ε, ο κυρκαδιανός ρυθμός των ανθρώπων ακολουθεί τα άστρα στην πραγματικότητα, όπου είναι ο ήλιος, αυτό θέλουμε κι εμείς, οπότε αυτά τα βραβεία, ξέρετε, δεν δίνονται έτσι χωρίς λόγο, αλλά ε, σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν καταλήξει σε επιτεύγματα επιστημονικά. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συζητάμε λοιπόν ε, την πρόταση της Κομισιόν. Το 2015 είχαμε φοβερά προβλήματα εδώ στην Τραν, στην Ένβη. Εμένα με εκπλήσει ακόμη και το γεγονός ότι καταλήξαμε να το συζητούμε αυτό το θέμα. Έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος, γιατί στην αρχή της συζήτησης αντιμετωπίσαμε σοβαρότατα προβλήματα. Όταν στην Φιλανδία θεσπίστηκε για πρώτη φορά η θερινή ώρα, ήταν όταν είχα γεννήσει το πρώτο μου παιδί και το θυμάμαι για αυτόν τον λόγο πάρα πολύ καλά. Ε, θυμάμαι ότι το επιχείρημα ήταν ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερη ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας. Ε, ότι ε, πρέπει να ε, εμείνουμε σε αυτήν την ε, θέση και όχι να θεσπίσουμε μεταβατικές περιόδους μέχρι το 2021. Και το Κοινοβουλίο έχει να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο εδώ. Το ίδιο βεβαίως και τα κράτη-μέλη τα οποία θα κληθούν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις. Το είπε και ο κύριος Σφόμποντα ότι στην, στο επίκεντρο της προσοχής μας πρέπει να είναι η υγεία του ανθρώπου, η δημόσια υγεία. Αυτό άλλωστε μα λένε και οι εμπειρογνώμονε. Θα έχουμε σήμερα και την ευκαιρία να ακούσουμε σχετικέ πληροφορίε και από εκεί και πέρα μπορούμε και να δούμε πώ θα προχωρήσει η συζήτηση αυτή και τι είδου αποφάσει θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη. Πάντω έχει δίκιο η κυρία Μάισνερ. Στη Ρωσία σήμερα πια δεν αλλάζει η ώρα. Υπάρχει η θερινή ώρα η οποία είναι η κανονική ώρα πλέον, ακριβώς γιατί διαπιστώθηκε ότι η συνεχής αλλαγή της ώρας ανεξάμεινο δημιουργούσε προβλήματα διαφόρων ειδών. Και τέλος θέλω να πω ότι μέσω της κατάργησης της οδηγίας κάποιες χώρες μπορεί εν τέλει να καταλήξουν να αλλάξουν την κανονική τους ώρα. Γιατί η Ισπανία, η Φιλανδία μπορεί κάποιο να πει ότι βρίσκονται, και στη λάθο ε, ώρα, ε, ζώνη ώρα. Οπότε μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για να γίνουν αλλαγέ ε, ε βελτιωτικέ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε στους ομιλητές, ε, τους μεμονωμένους, γιατί έχουμε λίγο, και λίγο γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει, ο κ. Ντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αρχίζουμε να αναλύουμε το θέμα αυτό. Πραγματικά διχάζει πολύ τον κόσμο. Εάν κοιτάξουμε ότι τα συμφέροντα των κρατών μελών δεν είναι τα ίδια, ε, προφανώς έχουν να κάνουν και με τη γεωγραφική τους θέση. Η γεωγραφική θέση ήταν καθοριστική και για το πακέτο κινητικότητας και πραγματικά με προξενεί ε, έκπληξη η παρατήρηση του συναδέλφου για το πακέτο κινητικότητα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να κάνει προτάσει που να μην διχάζουν, αλλά να ε, οδηγούν σε σύγκληση άποψεων την Ευρώπη. Διότι έχουμε ήδη το πακέτο κινητικότητα Τώρα ε, έχουμε ένα νέο μήλο της διχόνης μεταξύ των ε, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Η δουλειά της εισηγήτριας για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή, όμως δυστυχώς θα επιφέρει χάος στην Ευρώπη. Στην πράξη τι θα γίνει ας πούμε στη Γαλλία, πώς θα συντονιστεί η Γαλλία με τις υπόλοιπες χώρες. Ε, δεν αρκεί λοιπόν απλώς μια αλλαγή της οδηγίας για να αλλάξει μια παγιωμένη κατάσταση. Ποιο είναι αυτό το τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Διότι οι διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, δίνουν και διαφορετικές ερμηνείες. Αν ακούσουμε τι συζητιέται για την υγεία, για την οδική ασφάλεια κτλ., οι απόψει δίστανται. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπω τελικά η πρόταση αυτή δεν είναι και τόσο ε, απαραίτητη και ίσως η τωρινή λύση ε, που προτείνεται με την ηλιακή ώρα και την θερινή να είναι η λιγότερο χειρότερη, για να το πω έτσι από τις διάφορες συμβαστικές λύσεις που έχουμε. Μην ε, μπερδέψουμε τα πράγματα περισσότερο στην Ευρώπη. Επίσης, θα έλεγα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της. Εγώ θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Διότι δεν πρέπει να ε, ε, δώσουμε περισσότερη νομιμοποίηση σε μια τέτοια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα ήταν να αναβληθεί ή μάλλον να αναπενθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, δεχτούμε την εξοπλισμένη λύση που ήδη έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Κόχ. Ευχαριστώ Άρρωστοι δεν γινόμαστε ούτε λόγω τη θερινή ούτε λόγω τη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή από τη μία στην άλλη είναι αυτή που προκαλεί τα προβλήματα. 20% περίπου των Ευρωπαίων πλήττονται από αυτή την αλλαγή και θέλουν την κατάργησή τη. 80% των Ευρωπαίων από την άλλη πλευρά δεν έχουν κανένα πρόβλημα με του σημερινού κανόνε, αλλά δεν θα είχαν αντίρρηση και στο να καταργηθεί αυτή η αλλαγή. Εγώ λοιπόν θέλω 100% των Ευρωπαίων να είναι ευχαριστημένοι με το τι κάνουμε με την ώρα μα, γι' αυτό και υποστηρίζω την πρόταση τη Monsieur Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο. Δύο παρατηρήσεις, πρόεδρε. Πρώτα, μία ανάντη και μία κατάντη. Καταρχάς, τα μειονεκτήματα ή τα πλεονεκτήματα της αλλαγής της ώρας, τέλος πάντων της χειμερινής της θερινής ώρας, είναι τελείως ποικιλόμορφα, ε, αντικρουόμενα μεταξύ τους και αντιφατικά. Ο καθένα έχει τι δικέ του ευαισθησίε και αναλόγω με αυτέ μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ τη μια ή τη άλλη λύση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να τοποθετηθεί κανεί οριστικά επί του θέματο. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, λε και είναι το μεγαλύτερο τη πρόβλημα. Ενώ στην ουσία είναι μια λεπτομέρεια. Επίσης, στον κανονισμό δεν φαίνεται να υπάρχει καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει τώρα και τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή θα προκύψει πλήρη αταξία στο τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Μια αταξία που θα έχει και σοβαρέ συνέπειε για την εσωτερική αγορά. Για τι μεταφορέ λόγου χάρη. Και όχι μόνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ήταν πραγματικά χρήσιμη και υποδοματική η πρόβλεψη αυτή τη πρόταση τώρα. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά όμω. Είναι η στιγμή να υποβληθεί αυτή η πρόταση. Και μάλιστα χωρί καμία επικοδομητική συνέχεια για το τι θα γίνει αν υλοποιηθεί. Εντάξει, λέμε να διαλέγουν οι χώρε. Η θερινή όμω ώρα δεν είναι η ίδια στη Φιλανδία και στην Πορτογαλία. Δεν έχει τι ίδιε συνέπειε. Είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε, εάν δεν υπάρξει προσπάθεια ομογενειοποίηση, θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από ότι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα μπλοκαριστεί η πρόταση στο ε, Συμβούλιο. Ε, και τώρα θα ταχθώ υπέρ τη πρόταση του κυρίου Βαντεγκάμπ ε, διότι δεν είναι, θέλω να συμφωνήσω μαζί του απλώ επειδή θα φύγει από την ομάδα, αλλά πραγματικά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, να μην δεχτούμε μια πρόταση που δεν έχει καμιά δουλειά εδώ πέρα. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο, λέει πρόεδρος, ε, είναι δημοκρατικό όμως το αίτημα. Εδώ και χρόνια μας ε, στέλνουν επιστολές οι Ευρωπαίοι πολίτες και μας λένε εσείς πολιτικοί θύνοντες δεν θα προβλέψετε κάτι στην ημερησία διάταξη, τίποτα δεν θα συζητήσετε το θέμα αυτό. Να λοιπόν που τώρα το καλό μας Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προέβλεψαν το θέμα αυτό με μια ψηφοφορία ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τερματίσει την αλλαγή τη ώρα. Διαβουλεύσει γίνανε. Τώρα, συμφωνούμε ή όχι, οι διαβουλεύσει αυτέ ήταν ε, μεγάλη κλίμακα. Περίπου 5 εκατομμύρια πολίτε μόνο φέτο το καλοκαίρι. και κάποιοι έρχονται και λένε πολύ ξεκάθαρα ότι φτάνει, βαρεθήκαμε την αλλαγή. Τώρα ποια θα είναι η θέση διατησίας που θα πρέπει να λάβει το Συμβούλιο, θα έλεγα οι Υπουργοί Μεταφορών κυρίω θα πρέπει να αποφασίσουν επί Ρωμανική Προεδρία. Τότε θα συζητήσουν. Θα του θέσουμε το ερώτημα απευθεία. Διότι δεν θεωρώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αυτή την απόφαση και να καταλήξει σε συμπέρασμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω μπορεί να μα πει ότι κάποια πράγματα φαίνεται ότι τα. Ε, σας έφεραν πρωτοτελεσμένο με την ε, αποστολή αυτής της πρότασης και την, ε, τον δημοκρατικό αναβρασμό βρέθηκε και μια πρόταση που δεν προβλεπόταν ως προτεραιότητα στην ατζέντα σα. Ο κύριος Άρογκαρτ, λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται με την πρόταση διότι είπαμε να τερματιστεί η αλλαγή της ώρας, πολύ το θέλουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα το παραπέμπουμε στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι θα γίνει Μήπω πρέπει να γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσει με του πολίτε στην κάθε μια χώρα ξεχωριστά και μετά να συζητήσουμε και με του κρατικού φορεί και μετά να δούμε και με του ε, υπουργού μεταφορών, γιατί το είπαν και η κυρία Μπιλμπάο και η συγκεκριά μα και σωστά. Προσοχή, υπάρχουν τομεί που χρειάζονται χρόνο, όπω η αεροπλοεία, οι μεταφορέ. Εσεί λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πείτε μα πώ θα το ε, καλύψετε τον το αυτό με τις ανάγκες του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και καλό σα απόγευμα και στην εισηγήτρια και στους και εισηγητές επίσης καλησπέρα. Ευχαριστώ την κυρία Ολουσκοφ για τη δουλειά τη Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών στην ώρα και τις τροπολογίες που έχουν ήδη υποβληθεί. Ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ και την πολύ καλή παρουσίαση ε, της εκπροσώπου της κυρίας Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνολική στήριξη για την πρότασή μας να πάυσει η ετήσια αλλαγή ώρα μεταξύ θηρινή και χειμερινής. Με χαρά σημειώνω ότι συμφωνείτε στην ανάγκη να διατηρήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση στις αποκές αλλαγές ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή μας, είναι κρίσιμη σημασία για να είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργεί εύρυθμα η εσωτερική αγορά. Επίσης, σημειώνω ότι υποβλήθηκαν τροπολογίες για την έγκαιρη θέση σε ισχύ και υλοποίηση της πρότασης αυτής στην τελική της εκδοχή, δηλαδή όπως θα επικοινοποιήσει την οδηγία. Εμείς προτείνουμε ήδη φέτος να πάυσουν οι αλλαγές, αλλά είχαμε βασιστεί στην ε, υπόθεση ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία οι συνομοθέτες πριν την ε, εκλογική διακοπή του Κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται αυτό τώρα δεν θα συμβεί, οπότε προβλέπουμε περισσότερο χρονικό περιθώριο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια για συγκεκριμένε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί, όπου ζητήθηκαν αποσαφηνήσει και όπου έχουν ε, αναφερθεί και κάποιε ανησυχίε. Τροπολογία 5. Προτείνεται η διαγραφή στην αιτιολογική σκέψη 6 της μνήας ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να αλλάξουν την ε, παγιωμένη ώρα τους ε, και να την αλλάζουν πάνω από μια φορά το χρόνο. Η συγγήτρια θεωρεί ότι θα είναι εξαίρεση όμω η ώρα παρά ο κανόνα. Αυτό ακριβώ θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή τη. Στόχο είναι να υπογραμμίσουμε ότι η πρόθεση του Ευρωπαίου Νομοθέτη είναι να αποφευθεί η πιθανότητα τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να αλλάζουν την ε, κλασική του ώρα κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο ας πούμε επανεισάγοντα την εποχική αλλαγή τη ώρας από το παραθυράκι. Θα ήταν κάτι επιζήμιο για την εσωτερική αγορά αυτό. Γι' αυτό λοιπόν συνηγορούμε θερμά υπέρ τη διατήρηση τη μνήμα πάνω από μια φορά ετησίω More than once every year. Επίσης, σημειώνω την πρόταση τη εισηγητρίας στην τροπολογία 6 και 8 για τι ιδεολογικές σκέψεις 7 και το άρθρο 1 όπου η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εξορισμού επιλογή θα πρέπει να είναι η χειμερινή ώρα ε, η οποία να ισχύει από το Γενάρη και Εάν κάποια κάτι μέλη το επιθυμούν, να αλλάξουμε τελευταία φορά προ τη θερινή το Μάρτιο. Εμεί στη δική μα πρόταση υποτείνουμε ω εξορισμού κανονική ώρα την θερινή και επιτρέπουμε το φθινόπωρο να γίνει αυτή η τελευταία αλλαγή από τα κάτι μέλη. Η πρότασή μα παραμένει. Τα κάτι μέλη θα πρέπει να κάνουν την τελική επιλογή τη μόνιμη ε, τυποποιημένη του τη ε, πάγια του. Η εισηγήτρια ζητά από τα κράτη-μέλη να ορίσουν και ένα εθνικό σημείο επαφής με την τροπολογία 7 και 8. Κατανοώ ότι η εισηγήτρια Το προτείνει αυτό για να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί ο συντονισμό των ταξιδιών κρατών μελών. Κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και εμεί και το συζητήσατε και εσεί μόλι τώρα. Ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θεωρούμε όμω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το διοικητικό άχθο που θα επιφέρει κάτι τέτοιο και να λάβουμε και υπόψη τι αρμοδιότητε των κρατών μελών, που είναι ένα σημαντικότατο θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μπορούν να ορίσουν την πάγια ώρα του και να μην παρέμβει ε, ενοχλητικά, κατά τρόπο ενοχλητικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στι αρμοδιότητε των κρατομελών. Η πρότασή μα ω πρωταρχικό στόχο έχει τι εποχικέ αλλαγέ τη ώρα. Τέλο, με την τροπολογία 9 και 10, η συγγήτρια προτείνει ε, μια ελαφρώς διαφορετική συλλογιστική ως προς την ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών όταν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να αλλάξουν την παγιωμένη του ώρα και περάσουν από τη μία, χρονο, ε, τη μία ζώνη, την ζώνη ώρας προς την άλλη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως υπάρξει περισσότερο κόστος σε διοικητικό άχθος για τις εθνικές αρχές με την πρόταση αυτή. Η συγκεκριτή επίσης προτείνει να παραταθεί η ε, προθεσμία για την κοινοποίηση από 6 σε 8 μήνες. Καταλαβαίνω ότι η παράταση αυτή θέλει να επιτρέψει σε περισσότερους φορείς να προλάβουν. Να προετοιμαστούν δηλαδή και να είναι έτοιμοι για την αλλαγή. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε εδώ τη σωστή προσέγγιση ώστε και τα κατημέλη και το γενικό κοινό, δηλαδή όλοι οι πολίτες, να ενημερωθούν εγκαίρως και επαρκώς για τις ε, επερχόμενες αλλαγές με το λιγότερο δυνατό άχθος. Επίση, οι η θα πρέπει να λάβει υπόψη και τι απόψει και των άλλων ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ακούσαμε τι απόψει κάποιων σχεδόν εισηγητών τώρα το απόγευμα, οπότε δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τις δικέ του προτάσει, καθότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ελπίζω πάντω ότι η συζήτηση στην Επιτροπή σα θα οδηγήσει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα και σα ευχαριστώ και πάλι για την δουλειά σα. Ε, αν υπομονούμε για την τελική εκδοχή τη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σα κυρία Χέντ. Σας ξαναδίνω το λόγο για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ εκ μέρους της εισηγητρίας της Μαρίτα Ούλσκοφ. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρεμβάσει τους. Τα σημειώνουμε με μεγάλη προσοχή και θα φροντίσουμε να τα παραπέμψουμε στην εισηγήτρια. Έχω την εντύπωση ότι τα σχόλια που έγιναν και τα θέματα που τέθηκαν είναι θέματα που ήδη έχει αναφέρει στην έκθεση της και η κυρία Ολσκοφ. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη συνεργασία. Σα ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών προβλέπεται για τι 28 Ιανουαρίου το μεσημέρι στι 12. Και τώρα συνεχίζουμε με τη μεγάλη μας ακρόαση για το θέμα αυτό, για την πρόταση αυτή οδηγίας. Τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και ε, κατάργηση της οδηγίας 2084. Προσκαλώ τους εμπειρογνώμονε μας να ανέβουν στο Προεδρείο για να μπορέσω και να σας συστησω Allez, nous commençons. Ξεκινάμε και σας παρουσιάζω τους ε, ομιλητές. Τον καθηγητή Μπορκόφσκι. Καλώς ήρθατε. Στην ε, συνεδρίασή μας είστε, αντι... και υπεύθυνο για τις πολιτικές μεταφορών και οικονομίες στο Πανεπιστημίο του Γκτάνσκ στην Πολωνία. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Ο Δόκτωρ Κίραν Σάρμα, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Εσείς ε, εστιάζετε στις συνέπειες ε, της ε, πάυσης των αλλαγών ωραρίου με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια και είστε μέλος του Πανεπιστημίου του Galway στην Ιρλανδία. Έχουμε επίσης μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλευτικού Ινστιτούτου, τον κύριο Άντριου Τζάρβις, εσείς περισσότερο ασχολείστε με τον αντίκτυπο που θα έχει κάτι τέτοιο στην εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτού του θέματος μας ορκίστηκαν ότι θα έχουμε τεράστιες οικονομίες. Και έχουμε τέλος και τον κύριο Καστροβιέχο, Καλώς ορίσατε. Εσείς ε, μας έρχεστε από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα και είστε ο ειδικό για όλα τα θέματα τα ιατρικά, φυσιολογία και υγεία δηλαδή ανθρώπων και ζώων, ποιες είναι οι συνέπειες. Ωραία, λοιπόν, σας σύστησα όλους. Θα είμαι πολύ αυστηρή όμως μαζί σας, διότι δεν έχουμε το χρόνο. Όμως, συνάδελφοι, πιστεύω πως αυτή η ακρόαση είναι σημαντική. Γι' αυτό το θέμα της αλλαγής ωραρίου. Σήμερα θέλουμε λοιπόν να συλλέξουμε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διάφορες επιλογές και την πρακτική τους εφαρμογή. Γι' αυτό αποφασίσαμε η Επιτροπή Μεταφορών να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο για αυτό το θέμα ώστε ακριβώς να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όπως βλέπετε και ακόμα κι αν ε, το σημερινό θέμα ε, δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο, το Ευρωπαϊκό Επιτροπή ε, Κοινοβούλιο και Επιτροπή που συμφωνούμε σε αυτό το θέμα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας μετά από την ε, δημόσια διαβούλευση και να θυμίσω ότι 80% από τα 5 σχεδόν εκατομμύρια που ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση είπαν ναι θέλουμε να σταματήσουν οι αλλαγές της ώρας. Άρα λοιπόν Βασική μας μέρημνα ήταν η οικονομία ενέργειας. Είδαμε όμως ότι περισσότερες μελέτες έχουν αναπτυχθεί και δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στην ασφάλεια. Για παράδειγμα, στην Γαλλία υπάρχει μια έχμη ατυχημάτων συν 40% όταν γίνεται η αλλαγή ώρα από τη θερινή στην χειμερινή ώρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει οι μελέτες για την οδική ασφάλεια. Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία θέλουμε στη διαθεσή μας για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Και με χαρά σας υποδέχομαι ε, κύριοι εμπειρογνώμονες ώστε να μας ε, παρουσιάσετε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα των μελετών σας για αυτό το μεγάλο θέμα. Ποιος θα είναι λοιπόν ο αντίκτυπος μιας τέτοιας αλλαγής για τις ε, ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων στην υγεία, ε, στην οικονομία. Είστε λοιπόν ευπρόσδεκτοι, έχετε περιορισμένο χρόνο αγόρευσης, το ξέρω ότι αυτό μπορεί να σας προβληματίζει. Έχετε λοιπόν 8 λεπτά έκαστος ώστε να ξεκινήσει η μεγάλη συζήτηση με τους βουλευτές μας. Και κύριε Μπορκόφσκι ξεκινάμε με σας που έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Okay, thank you uh, for allowing me to share with you some of Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω την έρευνά μου που βασίζεται στην διαβούλευση που είχαμε με εκπροσώπους του κλάδου. Με τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και την αεροπορία. Να ξεκινήσω με τις οδικές μεταφορές. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που συλλέξαμε. Γιατί αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι ότι περιμένετε να υπάρχουν σοβαρές θετικές αλλαγές. Ε, για τις επιχειρήσεις μάλλον αδιάφορη είναι μια τέτοια αλλαγή όμως πρέπει να σας πω. Οι εταιρείε λοιπόν περιμένουν να κάνουν κάποιες πολύ μικρές εξοικονομήσεις ε, δαπανών, ιδίως αυτό μάλιστα αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, από τις δευτερογενείς δηλαδή οδικές μεταφορές που έχουν συνήθως το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς είναι ο χρόνος ανάπαυσης των οδηγών. Από αυτή την άποψη επειδή η αλλαγή της ώρας γίνεται κάθε φορά το, το Σαββατοκύριακο δεν θα αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα για τις επιχειρήσεις και του, του κλάδου των οδικών μεταφορών. Λίγες εταιρείε δηλαδή θα επηρεαστούν. Αυτό που φοβούνται οι εταιρείε πραγματικά είναι ε, αν θα υπάρξει μια αντικατάσταση της σας κατάστασης με μια μη συντονισμένη κατάσταση και μια κατάσταση όπου το κάθε κράτος μέλος ε, θα λαμβάνει τη δική του ε, απόφαση. Ακόμα και εναρμονισμένη πάντως να είναι αυτή η κίνηση, ε, δεν περιμένουν οι εταιρείε να έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές, ούτε εξοικονομήσεις, εκτός από ίσως κάποιες βελτιώσεις στο συντονισμό των βαρδιών εργασίας. Επίσης περιμένετε, αναμένεται μάλιστα να υπάρξουν και κάποιες επιπλέον δαπάνες, ένα ε, επιπλέον κόστας, κόστος ε, από μιας τέτοιας κατάργησης. Στις ιδοδρομικές μεταφορές τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί εκεί πράγματι το χρονολόγιο πρόγραμμα των, ε, των δρομολογίων θα επηρεαστεί. Παρ' όλα αυτά μιλάμε μόλις για το 5% των δρομολογίων που γίνονται ε, και τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή της θερινής ώρας. Επειδή κάποιο τρένο μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από ότι ε, μάλλον να φτάσει στον προορισμό του νωρίτερα ή αργότερα αντίστοιχα ανάλογα με το ποια αλλαγή γίνεται. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, ε, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή στις υποδομές των σιδηροδρομικών γραμμών ε, ούτε όσον αφορά τις εξοικονομήσεις γιατί το, τα φώτα τα ανάβουν έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από το τι ώρα είναι για τον ε, εποχιακό ε, προγραμματισμό ούτε αυτός θα επηρεαστεί γιατί δεν βασίζεται ούτε επηρεάζεται από, τις, από την θερινή ή τη χειμερινή ώρα ο συγκεκριμένο. Τα δρομολόγια παραμένουν τα ίδια. Ούτε αυτό λοιπόν θα έχει μεγάλες α, ε, επιπτώσεις γιατί όλες και οι δευτερεύουσες υπηρεσίες αποβίβασης, επιβίβασης έτσι και αλλιώς προσφέρονται ανεξαρτήτως της αλλαγής. Βεβαίως θα υπάρχουν κάποια ωφέλη για τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Αυτοί θα ωφεληθούν βασικά. Αυτοί που δεν, που δεν τους, αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι εταιρείε. Υπάρχουν όμως κάποιες ε, ε, ε, ε υπηρεσίες αποβίβασης που παρέχονται από τοπικούς περιφερειακούς φορείς οι οποίοι δεν συντονίζονται πάντοτε ε, με, τα, με τις στου εταιρείες ε, στους πελάτες θα υπάρξει ένα μικρό όφελος. Ωστόσο Για να, για να αποφεύγονται δηλαδή οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ε, παροχή υπηρεσίας τις ημέρες που αλλάζει η ώρα αεροπορικές εταιρείες. Εκεί δεν υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές που να αναμένονται γιατί και εκεί έτσι και έτσι παγκόσμιο είναι το, χρονολόγιο, το ορολόγιο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται και τα προγράμματα με βάση αυτό ε, καταρτίζονται. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν αναμένεται να υπάρξουν ούτε σημαντικές εξοικονομήσεις καυσίμων ή ενέργειας μια ανακατανομή θα γίνει στην ουσία των ορολόγιων προγραμμάτων πτήσεων ε, και ε, μπορεί μάλιστα να υπάρξει κάποιο κόστος λόγω της προσαρμογής που θα χρειαστεί να γίνει. ο αναπρογραμματισμός ε, βεβαίως θα διευκολυνθεί αν δεν υπάρχουν ε, περιφερειακές και τοπικές αλλαγές της ώρας. Ούτε, ούτε αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα με τις, ε, ε, ε, με τις πτήσεις τις διαδοχικές. Ε, και εδώ ε, αν υπάρξει κάποιο όφελος αυτό αναμένεται να υπάρξει στην πλευρά των πελατών, των ταξιδιωτών δηλαδή. Ποια είναι τα μεγαλύτερα θέματα λοιπόν και ποιες είναι οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις που μπορεί να γίνουν αεροδρόμια και διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων. Εδώ μιλάμε για το βασικό θέμα. Κάθε εποχική αλλαγή σημαίνει ότι γίνεται μια ανακατανομή, αναδιανομή των χρονοθυρίδων μεταξύ των αεροπορικών εταιριών. Αυτό βέβαια, αφορά κυρίως τα μεγάλα αεροδρόμια έντονης κυκλοφορίας, δεν αφορά τα τοπικά ή τα περιφερειακά ε, αεροδρόμια, όπου υπάρχουν διαθέσιμες χρονοθυρίδες πάντοτε. Μιλάμε για τα μεγάλα αεροδρόμια και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτοί πράγματι θα ωφεληθούν σημαντικά. Και ισχυρίζονται οι εταιρείες του κλάδου ότι σε περίπτωση που καταργηθεί η αλλαγή της ε, στη θερινή ώρα θα γίνει μια μεγάλη ανακατανομή η οποία πράγματι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κατανομή των χρονοθυρίδων. Και πάλι εδώ όμως ζητούμενο είναι να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση, Αυτό μας λένε. Ε, άρα, με δύο λόγια, ο κλάδος δεν αντιτίθεται, υποστηρίζει αυτήν την αλλαγή που προτείνει η Κομισιόν. Μικρές μικρά είναι τα ωφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν. Δεν θα υπάρξει, ε, ταυτόχρονα θα υπάρξει μικρό, ε, μια μικρή αύξηση του κόστους για τη διαχείριση και τη λειτουργία των υποδομών. Θα υπάρξουν όμως κάποια μικρά πάλι ωφέλη για τους επιβάτες. Αυτά. Κύριε Σάρμα. Um, Θα σας δώσω το πλαίσιο της σημερινής μου παρουσίασης. Ε, πρώτο σημείο είναι ότι η πρόταση για την πάυση των ε, αλλαγών ώρας δείχνει ότι όταν έχουμε μετακινήσεις σε περισσότερες ε, ε, λόγω της αλλαγής του φωτός θα έχουμε κέρδος στην ενέργεια. Ε, υπάρχουν πολλές ε, επιπτώσεις και το φως είναι, και η ορατότητα είναι μία από τις κεντρικές επιπτώσεις. Το δεύτερο είναι ότι η παρουσίασή μου έχει να κάνει με το χρόνο και το φως και αυτό διαφέρει ανάλογα με το μήκος και το πλάτος όπου βρίσκεται το κάθε μέρος. Έχουμε διαφορές ευδέ και κερικές. Επιπλέον έχουμε διαφορετικό αντίκτυπο στα διάφορα μήκη και πλάτη, ε, ιδιαίτερα ιδιαίτερα με μεταβλητές καθώς απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό. Ε, Τέλος να σας πω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μετακίνηση, μάλλον ότι η αλλαγή του φωτός προς το πρωινό ή προς το βράδυ ε, έχει να κάνει με το πότε χρησιμοποιεί κανείς τους δρόμους. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πότε πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ας πούμε, ε, πώς μπορεί να επηρεαστούν ε, οι αγρότες εάν δημιουργήσουμε πιο σκοτεινά πρωινά, γιατί περί αυτού πρόκειται σε ορισμένες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα όμως ε, έχουν, ε, η δική μου εισήγηση μιλά ε, για το ότι αν μετακινηθούμε προμονήμως προς τη θερινή ώρα μπορεί να έχει αυτό θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το να μετακινηθεί περισσότερη ορατότητα προς το βραδινές ώρες ε, μπορεί αυτό να σώσει πολλές ζωές. Είναι μια ε, υπόθεση μετακίνησης της ορατότητας και του φωτός. Η μόνη συνεπής, το μόνο συνεπές επιχείρημα σε σχέση με την οδική ασφάλεια εστιάζεται στην μόνιμη μετακίνηση προς τη θερινή ώρα και άρα στα φωτεινότερα βράδια ή απογεύματα. Με βάση αυτή την υπόθεση λοιπόν θα σας μιλήσω. Εδώ βασίζομαι σε 10 χρόνια στοιχείων ε, περί ατυχημάτων στην Ιρλανδία. Βλέπουμε δύο εχμές, η μία το πρωί είναι όταν ε, ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του και η άλλη το βράδυ η εχμή όταν ο κόσμος επιστρέφει πάλι. Ε, στο βαθμό που η εχμή η απογευματινή που είναι ψηλότερη από την πρωινή ε, θα είναι πιο φωτεινή με τη θερινή ε, ώρα, εάν μετακινηθούμε δηλαδή μονίμως προς τη θερινή ώρα, τότε θα έχουμε όντως θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Αυτή είναι η υπόθεση επί της οποίας ε, εγώ έχω δουλέψει. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με το βρετανικό πείραμα θερινής ώρας από το 68 μέχρι το 71, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε σταθερή την ώρα από το Μάρτιο του 68 μέχρι τον Οκτώβριο του 71. Και έχουμε στοιχεία για ατυχήματα, οδικά ατυχήματα και είδαμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος, βλέπουμε μάλλον ποιος ήταν ο αντίκτυπος. Η μελέτη δείχνει ότι αυξήθηκαν οι κίνδυνοι ατυχήματος το πρωί ε, ενώ μειώθηκαν για το απόγευμα βράδυ ε, οι περιπτώσεις ατυχημάτων και είχαμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές, αυτά είναι τα πορίσματα. Ωστόσο, εγώ ερμηνεύοντας αυτά τα πορίσματα θέλω να τονίσω τα εξής. Πρώτον, ότι αυτή η μελέτη είναι 50 ετών έχουν αλλάξει και η πυκνότητα της ε, κίνησης και ε, οι εξελίξεις στην ασφάλεια των ίδιων των αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Ε, είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτά τα πορίσματα σε όλες τις δικαιοδοσίες γιατί αλλάζει το φως στη διάφορα μήκη και πλάτη της γης. Και έπειτα, με αυτό το πείραμα, αυτό περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βρετανική κυβέρνηση πίστευε πως τελικά τα ωφέλη δεν ήταν επαρκή και έπειτα επειδή πίστευε ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο της Βόρειας Σκοτίας και επίση οι όσοι σηκώνονται νωρί είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο σκοτεινά πρωινά και η το ίδιο. Οπότε αυτή η μελέτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεν είναι παρκώς ε, αξιόπιστη. Τώρα, υπάρχουν διάφορες μελέτες όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις ε, το, της αλλαγής ώρας. Αυτό που έχει γίνει ας σε μία μελέτη είναι να μελετηθεί τι συμβαίνει ακριβώς μετά την αλλαγή, την θερινή και την χειμερινή και το 2017 εξετάσαμε 24 μελέτες που εξέταζαν τους κινδύνους ατυχήματος ε, τις ώρες, ε, τις, ε, τις μέρες μάλλον μετά την αλλαγή. Η αλλαγή στη θερινή ώρα οδηγεί σε αυξανόμενα ατυχήματα το πρωί και μείωση των ατυχημάτων το βράδυ. 12 εβδομάδες πριν και μετά κάθε αλλαγή. Έχουμε 12 σχετικέ μελέτες που οδήγησαν σε μικρέ που, που μάλλον έχουν ε, δείξει μικρότερες, ε, λιγότερα τυχήματα το πρωί, ίσω και λόγω τη μείωση όμω ε, τη κίνηση, επειδή κλείνουν τα σχολεία τη, η θερινή περίοδο. Και ε, Βεβαίω, στην αντίθετη περίπτωση, στην αλλαγή στο χειμερινό ωράριο, έχουμε και επιδείνωση του καιρού. Άρα υπάρχουν και διάφορες άλλες επιρροές. Οι, από αυτές τις μελέτες λοιπόν αρκετές έδειξαν ότι δεν υπήρχαν αλλαγή. Υπήρχε ωστόσο αρνητική επιρροή όσον αφορά την διάρκεια του ύπνου ε, στο θερινό ωράριο. Τώρα, η αλλαγή στο χειμερινό ωράριο σημαίνει μια επιπλέον ώρα ε, για το για, για, το βράδυ που σημαίνει όμως τελικά ε, πιο σκοτεινά βράδια και πιο φωτεινές, φωτεινά πρωινά. Από τις μελέτες αυτές ε, που έγιναν όσον αφορά την αλλαγή στο χειμερινό ωράριο πέντε από αυτές τις εκθέσεις δείχνουν αύξηση στα ατυχήματα και πέντε μείωση στα ατυχήματα και πέντε ε, έδειξαν ότι δεν υπήρχε αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το άσχημες χειρικές συνθήκες, διότι πρόκειται για τους χειμερινούς ε, μήνες ε, του χρόνου. Κάποια μικρά ωφέλη φαίνεται να υπήρξαν για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, αλλά δεν εξετάστηκε ο αντίκτυπος στα μικρά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο ε, το πρωί και γυρνούν ε, το βράδυ ενώ ακόμα έχει φως. Επίσης δεν εξετάστηκαν οι αγρότες. Τέλος λοιπόν, ποια είναι τα πορίσματά μου, ότι οι μελέτες αυτές έχουν ανάμεικτα αποτελέσματα, δεν ελέγχεται πάντοτε όλοι οι παράγοντες και δεν είναι σίγουρο ότι εφόσον μετακινηθεί η φωτεινότητα από το πρωί στο απόγευμα, ότι υπάρχουν δηλαδή σημαντικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Τώρα, ε, Εάν αποφασίσει η Επιτροπή σα λοιπόν τη μετακίνηση προς την θερινή ώρα, θα πρέπει να το αποφασίσει επί άλλη βάσης, όχι επί τη βάση τη οδικής ασφάλειας, διότι δεν έχουμε προβλέψιμα θετικά αποτελέσματα για τους χρήστε των δρόμων. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Να συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Τζάρβης κυρίως με ένα, μια ιδιαίτερη προσοχή στην ομιλία σας για την ενέργεια. Καλησπέρα σας. Ήμουν υπεύθυνο για μια μελέτη πριν από λίγα χρόνια, ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τι επιπτώσει τη θερινή ώρα εφόσον έπρεπε να είναι συγχρονισμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορούμε να δούμε τι επιπτώσει ορισμένα στον τομέα τη ενέργεια. Θα καταλαβαίνετε ότι ο πατέρας της θερινής ώρας, ο William Willett, είχε χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ότι η θερινή ώρα έχει μεγάλη σχέση με τις καταναλώσεις, ε, με την κατανάλωση στον τομέα της ενέργειας και μάλιστα είχε ξεκινήσει από την εξοικονόμηση ενέργειας στον Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 100 χρόνια η ιδέα αυτή. Η θερινή ώρα λοιπόν πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί ως ε, ένα μέσο για να εξοικονομηθεί υποτίθεται ενέργεια. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες δεν φαίνεται να είναι αμφισβητούμενες, όμως το ερώτημα είναι αν οι οικονομίες αυτές σήμερα έχουν κάποιο νόημα και αν θα χρειαστούν και στο μέλλον. Εάν δεν έχουμε πλέον τη θερινή ώρα, ίσως η κατανάλωση ενέργεια στην Ευρώπη να αυξηθεί και να αυξηθεί και η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα με απασχολήσει πιο πολύ στην παρουσίασή μου. Και συνεχίζοντα τι παρατηρήσει του συναδέλφου, θα πω ότι τα αποδεκτικά στοιχεία δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μια σειρά από μελέτε σε επίπεδο κρατών μελών, στην Ιταλία λόγω χάρη, την Γαλλία και την Ισπανία, όπω αναφέρονται και στη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται με αρκετή ασφάλεια ότι υπάρχουν κάποιες οικονομίες, όχι τεράστιες, αλλά σχετικές από την αλλαγή της ώρας προς το καλοκαίρι. Οι πανεπιστημιακές μελέτες ε, ανά τις χώρες δείχνουν ότι εκτιμήσεις επίσης υπάρχουν και με το σύνολο της Ευρώπης, τις 35 χώρες της, φαίνεται να υπάρχει ένας αντίκτυπος. Μεταξύ του 0 και του 2,5%. Βέβαια αυτό είναι απλώς ένα μοντέλο για τη μελέτη, δεν είναι καθαρή πραγματικότητα. Αλλά επηρεάζονται από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ε, τα δεδομένα. Και μάλιστα ε, δεν είναι μόνο το στοιχείο αυτό, αλλά ε, επηρεάζει γενικώ η γεωγραφική θέση Κάτι που δεν είμαστε σε θέση ακόμη να το εκτεμήσουμε ακριβώ. τώρα. Εάν δούμε λίγο περισσότερο σφαιρικά το θέμα, τα πράγματα είναι ακόμη πιο μπερδεμένα. Αν δούμε τι διεθνεί μελέτε, λόγω χάρη. Δεύτερη στον κατάλογό μου είναι μελέτη από τον Καναδά που δεν κατέληξε σε σαφή αποτελέσματα και μετά μια άλλη παγκόσμια μελέτη που βρήκε κάποια ωφέλη ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και την αλλαγή στη θερινή ώρα αλλά πολύ χαμηλή εξοικονόμηση. Εάν ξαναδούμε τώρα την ευρωπαϊκή μελέτη, μάλλον ήταν ε, λίγο πιο διαφωτιστική, έχοντας και κατά νου την ανάλυση που έγινε πριν από κάνα δύο χρόνια, από την υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας για τα τεχνολογικά θέματα. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου θα εξοικονομηθεί ενέργεια, όμως ε, θα μετατοπιστεί το πρόβλημα από κάποιες περιοχές σε κάποιες άλλες γεωγραφικά, λόγω των γεωγραφικών του συντεταγμένων, λόγω της γεωγραφικής θέσης και το, της χρονικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Τώρα, το θέμα είναι πώ διαμορφώνεται η ισορροπία δυνάμεων και απόψε μεταξύ των κατομελών στο Συμβούλιο και πώ θα έχει δει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι λόγω θερινής ώρα μειώθηκε κάπως η κατανάλωση ενέργειας. Αλλά αυτό φαινόταν από τη σφαιρικότερη προσέγγιση και όχι με τη λεπτομερή ε, ανάλυση σε μοντέλα. Πριν δηλαδή ρίξουμε να βλέπουμε το θέμα πιο καταλεπτό. Τώρα, στον τομέα τη ενέργεια, ένα βασικό μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρή υποστήριξη από τα αποτελέσματα τη πραγματικότητα για την τωρινή τακτική, αλλά από τα διασυνοριακά αποτελέσματα και τις πρακτικές, της εκπομπές αερίων φαίνεται να υπάρχει κάποια λογική στην αλλαγή της ώρας. Τώρα, το θέμα είναι πως μπορεί η κατανάλωση ενέργειας να επηρεάζεται από το φωτισμό και αν υπάρχει τέτοιου είδου εξοικονόμηση λόγω τη αλλαγή τη ώρα από το πέρασμα από τη χειμωνιάτικη ώρα στην καλοκαιρινή. Α υποθέσουμε δεν αλλάζει τίποτα. Είναι πιο αποτελεσματικό ο φωτισμό μα και έτσι ούτω ή άλλω έχουμε κάποια εξοικονόμηση ενέργεια. Όμω αρχίζει να λειτουργεί ο κλιματισμό περισσότερο. Άλλο επιστημονικό δεδομένο. Επίση κάτι που επενεχθήκατε στην συζήτησή σα νωρίτερα. Πώς θα καθορίσουμε το ποιε χώρε θα είναι στη θερινή ώρα, ποιες στη χειμερινή και πώς θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις εξοικονομίες στην ενέργεια. Δύσκολο, όχι μόνο προς τον άμεσο αντίκτυπο, αλλά και για να δούμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους λόγω των αλληλεπιδράσεων. Μπορεί δηλαδή ο κόσμος να μην πηγαίνει πια ποδήλατο, να κάνει ποδήλατο, αλλά να βλέπει τηλεόραση. Πάλι θα καταναλώνει ενέργεια. Δηλαδή είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πώ θα καταναλώνεται αυτή. Και προσπαθώντας να ολοκληρώσω την ε, σκέψη μου, δύο πράγματα που πρόκυψαν ξεκάθαρα στη μελέτη μας είναι ότι αν υπάρξει κάποια λύση αυτό που ελπίζουν οι ενδιαφερόμενοι ως προς το συγχρονισμό μεταξύ των κρατών για να μην υπάρξει χάος αυτό είναι σίγουρα κάτι που όλοι το επιθυμούν και μετά και η προσαρμογή του κόστους το αναφέρει και τελευταία μελέτη η δική μας υπηρεσία ελέγχου της κατάλληλης ενέργειας δεν έχει διασύνδεση στο διαδίκτυο αν δεν γίνει η αλλαγή της θερινής ώρας. Εγώ θα πρέπει να πάω να το κάνω αυτό με το χέρι αν ε, αποφασίσουμε να καταργήσουμε την θερινή ώρα. Οι λειτουργίες μας δηλαδή αυτές οι αυτόματες θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Δεν ήταν βέβαια αυτό ε, η ουσία τη δουλειά μα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μα παρήγγειλε αυτό το είδου τη μελέτη. Όμω είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα σκεφτούμε γιατί έχουν να κάνουν και με τον προγραμματισμό μα και με την καθημερινή διεξαγωγή των εργασιών μα. Ευχαριστώ. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σα Και τελευταίο μα προκεκλημένος ο κύριο Καστροβιέχο ο οποίος θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις και την καλή υγεία των πολιτών. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά. de cómo el cambio horario va a afectar a la salud. Ε, Πώς θα επηρεάσει η αλλαγή ωραρίου την ανθρώπινη υγεία. Καταρχάς να σας πω ότι όπως και τα ζωικά είδη ε, θα δείτε πώς επηρεάζονται από την αλλαγή των ωραρίων. Το ανθρώπινο «ον» αλλάζει τις δραστηριότητές του από την ημέρα στο απόγευμα και από το απόγευμα το βράδυ και αλλάζει επίσης και ο ρυθμός του ανάλογα με τις ε, ε, εποχές και αυτό διότι έχουμε ένα βιολογικό ρολόι σε κεντρικό επίπεδο και γνωρίζουμε πως ε, λειτουργεί χάρη στο Νόμπελ, στους ανθρώπους που κέρδισαν τον Νόμπελ το 2017 και έχει να κάνει με το ποσότητα του φωτός όσο και με τη διάρκεια του φωτός καθώς και με την ε, διαφορά ε, του είδους του φωτός. Λευκό το πρωί και ε, πορτοκαλί κόκκινο το βράδυ. Αυτό επηρεάζει την όρασή μας και με τη σειρά της εκείνη τα υπόλοιπα όργανα. Το σημαντικό είναι ότι έχουν ανακαλυφθεί πως όλα τα κύτταρα όλων των οργάνων ε, του οργανισμού μας έχουν ε, δικό τους βιολογικό ρολόι. Δηλαδή το ίδιο μοριακό και βιολογικό ρολόι. Έχουμε δισεκατομμύρια κύτταρα, δηλαδή έχουμε 30 δισεκατομμύρια κύτταρα και άρα 30 δισεκατομμύρια βιολογικά ρολόγια που λειτουργούν με ε, συντονισμένο τρόπο. Και η ώρα η κεντρική η συμπίπτει με την ώρα των περιφερειακών ρολογιών. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται η παραγωγή μελατονίνης η οποία μεταφέρεται μέσω του αίματος. Τις τρεις ε, το ξημερώματα έχεις περίπου τη μεγαλύτερη έκρηση και επηρεάζονται έτσι όλα τα περιφερειακά ρολόγια τα οποία συντονίζονται με το κεντρικό βιολογικό ρολόι. Όταν όμως αλλάζει η ώρα, η μηχανική, σημαίνει ότι θα πρέπει και το μοριακό μας ρολόι να αλλάξει ε, ώρα. Χρειάζεται όμως δύο-τρεις τουλάχιστον μέρες ώστε να συντονιστεί με την αλλαγή της ώρας. Άρα η μελατονίνη εκρίνεται όμως ε, κάποιες, ε, κάποια συγκεκριμένη ώρα και Άρα γίνεται έτσι μια, ένας αποσυγχρονισμός εσωτερικά που εκδηλώνεται με κάποιες φλεγμονές που μπορεί να οδηγήσουν σε δύρες λειτουργίες κεφαλικές, καρδιακές, μυϊκές, ακόμα και σε καρκίνο μπορεί να οδηγήσουν. Για να δούμε καλά πώς αλλάζουν όλα αυτά, έχουμε δύο παραδείγματα. Τώρα, αν εμείς ταξιδέψουμε από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο, έχουμε μια ώρα διαφορά. Όταν φτάνουμε στο Λονδίνο, λοιπόν, είμαστε, σηκωνόμαστε και ξαπλώνουμε μια ώρα αργότερα. Όμως, η ώρα της Ανατολής και της Δύσης είναι μια ώρα αργότερα. Άρα λοιπόν προχωρούμε προς την ίδια κατεύθυνση και άρα ο αποκοινωνικός εσωτερικός μας χρόνος που ορίζεται από το εσωτερικό μας ρολόι μας λέει πως είμαστε στην ώρα των Βρυξελών και προσαρμοζόμασταν γρήγορα. Αν όμως το φθινόπωρο κάνουμε το ίδιο, πάμε πίσω μια ώρα, πάμε δηλαδή συν δύο ώρες, κάνουμε το ίδιο όπως με το ταξίδι στο Λονδίνο. Όμως η ώρα ανατολής του ηλίου και δύσεις του ηλίου αυτό δεν αλλάζει γιατί δεν αλλάζουμε γεωγραφική θέση. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια δυσλειτουργία και η δυσκολία ε, ε, συγχρονισμού. Όλες αυτές οι μελέτες οδήγησαν σε μια σειρά κλινικών ε, παρατηρήσεων ε, πειραματικών και επιδημιολογικών και οδηγηθήκαμε στην έννοια του χρονικού κινδύνου. Σημαίνει δηλαδή υπάρχουν ε, περιστατικά νοσηρότητας ή και θανατηφόρα περιστατικά λόγω αυτών των σημαντικών αλλαγών. Μπορεί δηλαδή αυτές οι αλλαγές να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίε και σε παθολογίες. Πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα το εμφράγματος μυοκαρδίου που αυξάνεται ανάμεσα στο 5 και το 20% κάθε φορά που αλλάζει η ώρα κυρίως προς τη θερινή και επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και λιγότερο τους άνδρες μπορεί να έχουμε υψηλότερη αρτηριακή πίεση, χαμηλότερη χαμηλότερα λειτουργία το ανοσοποιητικό μας χρειάζεται να προσαρμοστεί ο εγκέφαλός μας ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε με το, την αλλαγή του ωραρίου. και να προσαρμοστεί και ο κερκαδιανός κύκλος. Έχουμε λοιπόν αύξηση αρνητικών ε, συμπτωμάτων, φλεγμονών, αλλεργιοπαθειών, ε, αρθρητικών και ένα σωρό άλλων παθήσεων. Και αυτό οφείλεται στον μη συγχρονισμό, τον μη, μη άμεσο συγχρονισμό του βιολογικού ωραρίου με την ε, ώρα, ε, την εξωτερική. Οι αλλαγέ του ωραρίου δεν οδηγούν σε καρκίνο, αλλά ε, επηρεάζουν ένα σωρό άλλους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε προδιάθεση για εμφάνιση καρκίνου. Το 2018 οι υπογράφοντες αυτής της εργασίας ε, του Ευρωπαϊκού ε, Περιοδικού Εσωτερικής Ιατρικής δείχνουν πώς οι αλλαγές ώρες μπορεί να επηρεάσουν τον κυρκαδιανό κύκλο και το βιολογικό μας ρολόι. Έχουν δημοσιευθεί μελέτες που αποδεικνύουν ε, τα αρνητικά επι... Ε, τις αρνητικές επιπτώσεις ε, των αλλαγών της ώρας στο κυρκαδιανό κύκλο. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές αποδείξεις ώστε να πούμε ότι οι αλλαγές της ώρας δεν θα πρέπει να διατηρηθούν και θα πρέπει να πάψουν. Τέλος να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιο θα ήταν το καλύτερο ωράριο σύμφωνα με το δικό μας βιολογικό ωράριο. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για την Ισπανία, αλλά μπορεί να το ε, δούμε και για οποιαδήποτε χώρα όπου βλέπουμε ότι η ποσότητα του φωτός ε, διαρκεί περισσότερο το βράδυ. Το πορτοκαλί είναι τα ωράρια εργασίας. Έχουν, υπάρχουν μικρές αλλαγές ε, στη διάρκεια των διαφόρων εποχών του χρόνου. Ενώ κάτω βλέπουμε ότι αν αυξηθεί λίγο το φως το πρωί και μειωθεί λίγο το βράδυ δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια των εποχών. Κάτω δεξιά βλέπουμε τον ώρα, κεντρική ώρα συν 2 έχουμε πολύ περισσότερο φως το βράδυ μέχρι αρκετά αργά το βράδυ και αυτό επηρεάζει πολύ δραστικά το βιολογικό μας ρολόι και παρεμποδίζει τους μηχανισμούς που θέτουν σε λειτουργία την ε, ανάπαυση. Βλέπουμε ότι το πρωί έχουμε περισσότερο φως το καλοκαίρι. Υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι. Ακριβώς και ε, με το φως το βράδυ που δεν φτάνει σε πολύ ε, ε, βραδινές ώρες. Άρα λοιπόν όσο λιγότερες είναι οι αλλαγές στις ώρες φωτεινότητας τόσο το καλύτερο ώστε να μην επηρεάζεται το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καστροβιέχο με την έμφαση που δώσατε στο θέματα της υγείας και θα αρχίσουμε αμέσως τη συζήτηση με τους συναδέλφους και ξεκινάμε με εσάς κύριε Βίμ Βαντερκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι θέλετε να δώσετε πρώτα το λόγο στους σκιώδεις συζητητές. Αλλά εντάξει. Πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσίασε η ισπανική μελέτη του κυρίου Καστροβιέχο. Δυστυχώς δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά το όνομα. Είναι πάντως ε, ε, πολύ σοβαρή η ετοιμιγορία, το πόρισμα στο οποίο καταλήγει η μελέτη αυτή. Έχω και να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Ε, σήμερα το πρωί ήρθατε στι Βρυξέλλε, φαντάζομαι αεροπορικό. Άρα σημαίνει ότι ξυπνήσατε και πάρα πολύ πρωί. Γιατί χρειάστηκε να φτάσετε έγκαιρα εδώ στη συνεδρίασή μα. Εσεί διατρέχετε τώρα τον κίνδυνο να ε, αναπτύξετε κάποια ασθένεια Ξέρετε όλοι όσοι είμαστε εδώ, κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια. Ερχόμαστε εδώ στι Βρυξέλλες, πάμε στο Στρασβούργο, πάμε στην Κίνα. Έχουμε δηλαδή καθο... έχουμε προγράμματα τα οποία είναι ε, μη προβλέψιμα πολλές φορές και πολύ διαφορετικά. Τι, τι, κινδύνους δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι διατρέχουμε λόγω αυτής τη αλλαγής που διατρέχουμε κάθε εβδομάδα εδώ στις εργασίες μας. Ευχαριστούμε κυρία Μπελμπάου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Από, να, να κάνω μια, ε, μια ερώτηση όσον αφορά την ε, επιχειρηματική πρόπτικη, ότι δηλαδή δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αντίθετα από ό,τι φαίνεται από την ε, προοπτική της υγείας, φαίνεται ότι αν λάβουμε μια τέτοια απόφαση θα έχει θετικό αντίκτυπο. Ερώτησή μου προς όλους. Με αυτή την έκθεση που έχουμε τώρα επιτάπητος, ποια είναι η σύσταση καθενός από εσά. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας για τις λεπτομερέστατες παρουσιάσεις τους. Εγώ έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Καστροβιέχο. Για όσα σχολιάσατε και από την σκοπιά της υγείας, υπάρχουν ε, γιατροί, βιολόγοι που ασχολούνται με τα θέματα της ώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και ιατρικές ενώσεις που έχουν τοποθετηθεί για τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν στην ανθρώπινη υγεία. Γνωρίζετε εσείς συγκεκριμένες αποφάσεις τέτοιων ενώσεων. Ευχαριστούμε κύριε Σάβαντα. Κυρία Κλούν. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας. Ε, νομίζω είναι σαφές η οδική ασφάλεια είναι ένα τεράστιο θέμα και το αναφέρατε σε κάποιε από τι μελέτε σα. Είναι δύσκολο βέβαια να καταγραφεί συγκεκριμένα. Α, το ίδιο και εξοικονόμηση ενέργεια. Ήταν από του βασικού λόγου που είχαν προταθεί αλλαγέ την ώρα όταν πρωτοπροβλέφθηκαν. Ε, ε, θα ήθελα λοιπόν για το σύνολο αυτού του τομέα και για το κατά πόσο η θερινή ώρα, δηλαδή η ώρα των Greenwich in 2 είναι καλύτερη για να έχουμε περισσότερο φως το βράδυ ας πούμε, αν είναι καλή ιδέα. για το βασικό κόστος και τις αλλαγές ένα εξάμεινο. Αλλαγή το Μάρτιο και τον Οκτώβριο από την πλευρά των επιχειρήσεων και από την πλευρά της ε, ευκολίας για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, του κατά πόσον η αλλαγή είναι πρόβλημα. Ευχαριστούμε κυρία Κλούν. Η κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή Μεταφορών που οργάνωσε αυτή την τόσο καλή ακρόαση. Εγώ εκπροσωπώ εδώ την Επιτροπή ΙΤΡΕ, είμαι μια τη εκεί. Και Έχω κάποια επικρατικά σχόλια, όπως ε, για τις μεταφορές. Τα ευρήματά τους ε, ε, δεν συμφωνούν απολύτως με τα δικά σας. Βλέπετε λοιπόν υπάρχει κάποια... να υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι καλύτερη μια ή άλλη λύση, γιατί δεν είδα πολλά να προκύπτουν για την ε, οδική ασφάλεια. Ε, στη Φιλανδία πολύ συχνά λένε ότι το θέμα της υγείας είναι σοβαρό για την οδήγηση. Ε, η υγεία ούτω ή άλλω. Αυτό ίσω είναι μια παράμετρο λοιπόν όχι απλώ για όσου οδηγούν, αλλά και για όσου οδηγούν διασυνοριακά. Εγώ, α πούμε, το έκανα σήμερα το πρωί. Είναι ίσω σχετικά απλό, αλλά δεν είναι και διασκεδαστικό. Και για την ενέργεια ήθελα να θέσω συγκεκριμένη ερώτηση. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο ενδεχόμενη ωφέλεια από την ε, ε, ε, από την πάυση, ε, τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας ή ίσως για το πώς θα θερμαίνονται ή θα ψύχονται τα σπίτια και οι χώροι. Ναι, δεν υπάρχουν άλλοι παραμένοντας. Θα κάνω και εγώ λοιπόν μια ερώτηση η οποία απευθύνεται περισσότερο στον κύριο Καστροβιέχο. Για τις ιατρικές συνέπειες, εάν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε και προσπαθήσατε να αποδείξετε, Η βασική όκληση είναι το θέμα της αλλαγής, της συστηματικής αλλαγής της ώρας για το βιολογικό ρολόι. Πέραν αυτού υπάρχουν συγκεκριμένες όμως για να προκρίνει κανείς ή τη θερινή ώρα ή τη χειμερινή ή αντιθέτως να τις δει διαφορετικά ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της κάθε χώρας. Είναι τελείως διαφορετική κάθε περίπτωση ε, και τελείως διαφορετική και γεωγραφική θέση των χωρών οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα. Θα απαντήσετε με τη σειρά με την οποία ε, εκφωνήσατε τις ομιλίες σας. Τρία-τέσσερα λεπτά απάντηση ο καθένας στις ερωτήσεις που τέθηκαν παρακαλώ. Και αν γίνεται τα πρακτικά σας συμπεράσματα να είναι μια συνθηματική διατύπωση εφόσον γίνεται. Ο κύριος Κοβόσκι που ξεκίνησε και την ε, ακρόαση. Λοιπόν, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για την πλευρά των επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις λοιπόν, για τις, για επιχειρήσεις του, του, του κλάδου των μεταφορών η αλλαγή αυτή δεν θα είναι σημαντική. Εκτός από τις ε, χρονοθυρίδες, όπως σας περιέγραψα. Αλλά όλοι ε, ε, όσοι μιλήσαν μαζί μας ήταν θετικοί. Είπαν εντάξει προχωρήστε. Με έναν αστερίσκο. Σας παρακαλούμε κάντε το συντονισμένα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν διάφορες ζώνες ώρας και κάθε κράτος μέλος να αλλάζει από μόνο του την ώρα του. Αν θέλετε να καταστρέψετε το σύστημα που έχετε αυτή τη στιγμή, καλώς, αλλά σας παρακαλώ κάντε το προς μια κατεύθυνση όπου όλοι θα κάνουν περίπου το ίδιο, με έναν συντονισμένο τρόπο. Um, on a position. Is that what we're... Για την πλευρά της οδικής ασφάλειας υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες κινδύνου που καθορίζουν τον κίνδυνο ατυχήματος που η μετατόπιση του φωτός ε, μία ώρα πριν ή δύο ώρα μετά δεν, δεν, δεν, υπάρχει, δεν έχει αποδειχθεί ότι πράγματι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα ατυχήματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ε, ούτε προς τη μία κατεύθυνση για τη διατήρηση της ε, θερινής ώρας, ούτε ότι θετικό, ε, θετικό αντίκτυπο θα είχε η κατάργηση αυτής της αλλαγής. Σημαντικό είναι οι συζητήσεις της Κομισιόν να μην προσπαθήσουν να εντάξουν το θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί δεν υπάρχουν έγκυρα ε, επιστημονικά στοιχεία. Ε, λόγω γεωγραφικού ε, πλάτους και μήκους υπάρχουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία τα που θα μπορούσαν στη μία ή στην άλλη χώρα να δείξουν ότι αυτή η αλλαγή μπορεί και τελικά να είναι ένας παράγοντας, όμως όταν βλέπουμε συνολικά τα στοιχεία για ολόκληρη την Ευρώπη δεν μπορεί να διαπιστωθεί με ασφάλεια και με ακρίβεια κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζάρβις. Ναι, θα προσπαθήσω να την απαντήσω σε μια-δυο ερωτήσει. Το τι θα προτείναμε συνολικά και μετά σε σχέση με την ενέργεια. Νομίζω η σφαιρική εικόνα είναι ότι αν το δει κανεί από την πλευρά των πολιτικών και της χάραξης πολιτικής υπάρχουν ε, λεπτομερείς μελέτες αντικτύπου που λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς παράγοντες. Η καλύτερη υπόθεση που μπορεί να κάνει κανεί είναι τα μελλοντικά σενάρια που θα κάνουν τα κράτη-μέλη ανάλογα με τη χρονική του ζώνη, τη ατράκτου και ε, το τι στάση θα υιοθετήσουν. Επίση, το κόστο για τι επιχειρήσει είναι σημαντικό. Η αλλαγή δι ετησίω είναι ένα θέμα για τι επιχειρήσει. Αυτό το κόστο μπορεί να υπολογιστεί. Οπότε πρέπει κανείς να σκεφτεί αν θα συζητήσει το κόστος της αλλαγή σε ένα καινούριο σύστημα. Επίσης, εάν υπήρχαν οι πόροι για να γίνει μια στατιστική μελέτη λεπτομερής σε επίπεδο μέλη μέλους και το τι κάνει ο καθένας πολίτης για να δούμε ποιες είναι οι δικές τους ανησυχίες, ποια είναι η δικιά τους ανάγκη, διότι ποιοτικά τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε δεν μα επιτρέπουν να το κρίνουμε αυτό με τι τόσο διαφορετικέ και αντικρώμενε απαντήσει. Και αν αυτά λοιπόν μπορούσαμε να τα συναθρήσουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται σε επίπεδο κράτου μέλου για την υγεία και την ε, εξοικονόμηση τη ενέργεια και το καθεξή, με ποιοτικού και ποσοτικού ε, παράγοντε. Ε, θα βλέπαμε ότι από όσου ασχολούνται με το εμπόριο τη ενέργεια και τι παρατηρήσει που έκαναν, αλλάζει η ζήτηση και η προσφορά για την ενέργεια στα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλάζει ανάλογα με την ε, α, ορολογική, ορολογική άτρακτο. Οπότε μπορεί ο συγχρονισμό να ε, επιφέρει μεγαλύτερο φόρτο για το δίκτυο. Σίγουρα θα αλλάξει η κατανομή της ζήτησης ανά τα κράτη-μέλη εάν το σύστημα μεταβληθεί. Ευχαριστούμε πολύ και για να ολοκληρώσουμε ο λόγος ξανά στον κύριο Καστροβιέχο. Bueno, eh, lo que usted comenta sobre... Mm, ναι, αυτό το θέμα του κατά πόσο επηρεάζεται κανείς αν ταξιδεύει πολύ με το αεροπλάνο είναι κάτι άσχετο. Γιατί για παράδειγμα υπάρχει πολλοί κόσμος που καπνίζει σαν φουγάρο αλλά δεν παθαίνει καρκίνο ενώ άλλοι που δεν καπνίζουν ποτέ παθαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ προβλήματα και άλλοι εγώ ας πούμε έκανα βάρδιες στο νοσοκομείο για χρόνια. Όλο το βράδυ έμενα ξάχρυπνο. Ε, το πρωί έκανα διαλέξει στο πανεπιστήμιο και άντεχα. Δεν έπαθα τίποτα. Όμω, άλλο είναι αν μπορεί να το κάνει, να αντέχει, και άλλο είναι αν μα επηρεάζει ή όχι. Εμεί είμαστε ζώα. Είμαστε ζώα και διεπόμαστε από νόμου που δεν είναι ακριβεί, δεν είναι φυσικοί ή μαθηματικά. Κάθε ζώο και κάθε ανθρώπινο όν μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα ότι η Κομισιόν πρέπει να νομοθετήσει όταν υπάρχουν παρατηρήσεις που λένε ότι οι σημερινοί νόμοι παράγουν, μάλλον οδηγούν σε προβλήματα υγείας. Κάποιες φορές υπάρχουν, ε, ε, ναι, δεν επηρεάζονται όλοι, ευτυχώς, αλλά αν λάβουμε υπόψη το ποσοστό ε, προβλημάτων υγείας, τότε είναι σημαντικό να ε, υπάρξει και σχετική νομοθεσία. Και μάλιστα αυτή είναι και η αρχή της προφύλαξης που ισχύει για οποιαδήποτε νομοθεσία. Αν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν βλάβη, θα πρέπει να το προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Τώρα, συγχρονισμός των ε, βιολογικών ε, ρολογιών. Πολλοί από τους υπογράφοντες ε, τις μελέτες αυτές είναι ειδικοί χρονοβιολόγοι από την Ισπανία, από την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, από τον Καναδά. Έχουμε συνευρεθεί, Θέλουμε μαζί να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε, ότι επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλαμε να συμβάλλουμε και να στηρίξουμε αυτά που συζητώνται εδώ. Υπάρχουν ε, βεβαίω δυσλειτουργίε και αυτό το παρατηρούμε πάρα πολύ καλά στα παιδιά. Γιατί υπάρχουν διαφορέ, υπάρχει μείωση προσοχή, μείωση τη μνήμη και τη δυνατότητα μάθηση τι ημέρε μετά την αλλαγή του ωραρίου. Και πάλι δεν επηρεάζονται όλα τα παιδιά. Μιλάμε για ένα ποσοστό. Βέβαια, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα και δείχνουν περισσότερο τις αλλαγές στις ικανότητές τους. Ποια θα ήταν η σύστασή μου τελικά. Καταρχάς, να, μην αλλάξουμε, να μην αλλάζουμε την ώρα. Δεύτερον, το βιολογικό μας ρολόι είναι έτοιμο για να δέχεται περισσότερο φως το πρωί και από τις 6-8 το βράδυ, το απόγευμα, να μειώνεται σιγά-σιγά η φωτεινότητα ε, προς ε, το πορτοκαλί και προς το κόκκινο ε, ε, να στρέφεται η φωτεινότητα. Ωστόσο, ε, έτσι το βιολογικό μας ρολόι μας ετοιμάζει για να αναπαυθούμε και να κοιμηθούμε. Το ωράριο είναι αυτό που, που ε, είδαμε και προηγουμένως ότι υπάρχουν διαφορές φωτός το πρωί και το βράδυ σε όλες τις εποχές. Αυτό κοιτάει το βιολογικό μας ρολόι για να λειτουργεί σωστά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Ε, είναι ακόμα πολλές οι απορίες παραμένουν αναπάντητες και τα ερωτηματικά. Το θέμα της οδικής ασφάλειας ας πούμε, όπου μας λέτε ότι η αλλαγή της ώρας δεν είναι σαφές αν θα επηρεάσει ή όχι. Συμφωνείτε όμως όλοι ότι αν σταματήσει και τερματιστεί η αλλαγή της ώρας και παραμείνουμε στη χειμερινή ή τη θερινή ώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνηθεί συντονισμός και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε ότι οι ανησυχίες και οι διαταραχές στην υγεία και στα παιδιά και στους ηλικιωμένους μπορεί να είναι σοβαρές. Και για τις οικονομήσεις στην ενέργεια και αυτό είναι επιχείρημα, διότι από το 1970 εξοικονόμηση στην ενέργεια γίνεται και λόγω των τεχνολογικών λύσεων. Δεν τα είπαμε αυτά. Α? Οι τεχνολογικές αλλαγέ έχουν επιτρέψει η εξοικονόμηση τη ενέργειας. Δεν είναι μόνο η αλλαγή τη ώρα. Το αποδείξατε άλλωστε με στοιχεία. Από 0,5% έως 2%. Πρέπει βεβαίως να πούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες είναι οι χώρες του 0,5% και ποιες είναι αυτές με το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ και 30-40 χρόνια πάντω που λειτουργεί το σύστημα αυτό δεν είναι τεράστιο αντίκτυπο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αποστήλαμε ένα σαφέ μήνυμα μετά το αίτημα των πολιτών. Είμαστε εδώ για να νομοθετήσουμε και νομίζω ότι το σύνολο των συμπερασμάτων σα επιτρέπουν να δούμε τα θέματα και τις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη προσοχή. Είστε πολύ εδώ στο Προεδρείο μαζί μου, κύριοι, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ Μπράβο σα. Χειροκροτήστε του, παρακαλώ. Σε τραβάει. Et je vais continuer mes, tra mes travaux. Allez-y, je vous laisse rejoindre la salle. Allez-y, merci à vous. Θα συνεχίσω τη συζήτησή μου. Θα σας αφήνω να επιστρέψετε στην αίθουσα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

Να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Απαλλαγές 2017. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Οργανισμοί. ΕΜΣΑ, ΕΑΣΑ, ΕΡΑ, ΣΕΖΑΡ και ΣΥΦΤΟΥΡΕΙΛ θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Βιν Βαντενκάμπ. Εκ μέρου του κυρίου Προύστ. Κύριε Λεοντίνη, θα πάρετε το λόγο μετά. Κύριε Βαντενκάμπ, εσεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Προύστ είχε αναλάβει την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο συνάδελφος Λεοντίνη τους υπόλοιπους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο σε, πρώτο, σε πρώτη φάση. Ε, ο κύριος Προύστ δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, οπότε απλώς θα σας διαβάσω την παρέμβασή του. Καταρχάς, θέλει να ευχαριστήσει θερμά του συνεργάτες της Επιτροπής Μεταφορών που τον βοήθησαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής για την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών σε ό,τι φορά το περιεχόμενο. Πρόκειται για απαλλαγή υπό την κλασική έννοια του όρου. Ο κύριος Προύστ δεν βλέπει φέτος να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν γίνει μια σειρά από αναλύσεις για τον προπολογισμό του 2017 και την εκτέλεσή του και η άποψη του κυρίου Προύστ, άρα και κατ' επέκταση του ΕΛΚ, είναι ότι όλα έχουν πάει καλώς. μια ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση, το ΣΕΦ, που ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό και είχε πολύ θετική απήχηση. Ε, ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη σχετική προσπάθεια για τα επόμενα χρόνια για να στηρίξει το ΣΥΕΦ, το οποίο αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί βέβαια σε τριμερή διάλογο Εκεί λοιπόν θεωρώ κύριο Πούστο ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα κίνητρα που δίδονται και να προσπαθήσουμε να τονώσουμε κι άλλο το ΣΕΦ, ώστε όλα τα μέλη των ε, Επιτροπών Τουρισμού και Μεταφορών να μπορέσουν να υπερψηφίσουν την πρόταση αυτή αύριο. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου του κυρίου Προύστ. Ευχαριστούμε κύριε Βιν Πεντακάμπ και τώρα ο λόγο στον κύριο Λεοντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως προς τις απαλλαγές για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2017 και όπως είπε και ο πρόεδρος Ντεκάμπ εγώ στι εκθέσει μου ασχολήθηκα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια τη Αεροπορία, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κοινή Επιχείρηση για την Ασφάλεια τη Αεροναυτιλία για τον ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ΣΕΖΑΡ και την κοινή επιχείρηση Shift to Rail. Έτσι ολοκληρώνεται το φάσμα των πέντε αυτών ευρωπαϊκών οργανισμών. Όπως όταν η διαδικασία απαλλαγής γίνεται και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ώστε να δούμε πώς δαπανήθηκαν δημόσια κονδύλια, τα οποία υποδιαιρέθηκαν μεταξύ των πέντε αυτών οργανισμών. Υποβλήθηκαν συνολικά 38 τροπολογίες, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα που θα έπρεπε να συζητήσουμε και συνολικά θεωρώ ότι οι τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί εμπλουτίζουν και φωτίζουν καλύτερα το κείμενο που έχω εκπονήσει εγώ ίδιος. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο επίπεδο της Επιτροπής. Προτείνω να δώσουμε την ε, απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς, έτσι όπως το αναφέρω και στα σχέδια εκθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Λεοντίνη. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κύριου Τιλίτσκα, ο οποίος ζητεί συγγνώμη που δεν είναι σήμερα εδώ, ε, είχε καθυστέρηση η πτήση του, βρίσκεται καθοδόν, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ για να πάρει το λόγο. Αν ε, ήταν εδώ, ε, το, τα μόνα πράγματα που θα είχε πει θα ήταν ε, ε, κάποια λόγια εκτίμησης για το έργο των εισηγητών. Οι τροπολογίες του αφορούσαν κάποια επουσιώδη θέματα, ιδίως όσον αφορά τον οργανισμό αεροπορίας και ελπίζει η έκθεση αυτή να τύχει της υποστήριξης όλων των μελών της Επιτροπής μας αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. αμέσως να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει κάτι να μας πει. Κυρία Μοντανιό, από την DG Move. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντες. Δύο κουβέντες για να εκφράσουμε και εμείς την ικανοποίησή μας για τη θέση που πήρατε. Και εμείς είδαμε ότι βήματα πρώτα έχουν γίνει σε πολλά επίπεδα Στου οργανισμού, απλώ να δώσω δύο διευκρινήσει σε σχέση με τι εκθέσει και ορισμένε τροπολογίε που υποβλήθηκαν επ' αυτών. Μας φάνηκαν σημαντικέ. Πολλέ τροπολογίε αφορούν την διακυβέρνηση, τη διεύθυνση δηλαδή των οργανισμών και κυρίω τα λογιστικά του και το οργανόγραμμά του. Είναι ένα σημείο επί του οποίου στράφηκε η προσοχή μα. Η κατάσταση τη ΕΜΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια τη Θάλασσα, ήδη πέρσι εξομαλύνθηκε της ΕΑΖΑ για την αεροπορία ήδη έχει ε, τακτοποιηθεί φέτο, δηλαδή θα ολοκληρωθεί η σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου την επόμενη φορά και το ίδιο και για την ε, ΣΕΖΑΡ. Τώρα, είδα πολλές τροπολογίες για τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών. Απλώς να διευκρινίσω για τις δυσκολίες που επισημάνατε κι εσείς για την ΕΑΖΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, μία περίπτωση ένα διαγωνισμό προσέκρουσε σε δυσχέρειε. Ε, για την πληροφορική. Όχι για όλε τι προμήθειε που οργανώθηκαν. Οπότε ο διαγωνισμό αυτό κράτησε πολλά χρόνια με ένα σύνολο προκοδότηση 15 εκατομμύρια. Αλλά δεν αναφέρεται στι αιτήσει αποφάσει χρηματοδότηση με το. Ε, ε, ετήσιο ποσό, το 5 εκατομμύρια προβλέπονται ετησίω. Γι' αυτό υπάρχει απόκληση μεταξύ του αριθμού που προβλέπεται στην περίοδο προγραμματισμού και την ετήσια απόφαση χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Εισηγητέ, θέλετε και πάλι το λόγο. Κύριε Βαντεγκάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να προσθέσω για την απαλλαγή Λάβαμε κάποιες τροπολογίες από τον κύριο Τελίτσκα, από τον κύριο Καπούτο, από τον κύριο Νταλούντε. Και η κυρία Αρνοτού επίσης υπέβαλε κάποιες τροπολογίες, ε, τροπολογίες που γίνονται δεκτές από τον κύριο Προύστ πλην τη τροπολογία 8 από τον κύριο Αρνοτή η οποία δεν γίνεται δεκτή από τον κύριο Προύστ. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Βαντενκάμπ. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουμε. Κύριε Λεοντίνη, θέλετε και εσείς το λόγο. Α, ωραία. Πολύ καλά. Είπαμε θα ψηφίσουμε αύριο στις 9. Α, λάθος. Τι λάθος. 10 ξεκινάμε. Μια ώρα παραπάνω θα, που θα κοιμηθείτε. Και τώρα κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης, διότι θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών για την ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους και τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ένα μικρό διαλυματάκι για να πάψει η μετάδοση στο διαδίκτυο και να φύγουν οι ε, παρήσακτοι του κοινού. Ε, οι βουλευτέ που είναι αρμόδιοι μπορούν να μείνουν. Αρχίστε να οδεύετε προς